ορίζεται η ημερήσια διάταξη για την τρέχουσα σύνοδο και περνώ στην έκθεση του κυρίου Μαρινέσκου, χαιρετίζοντα και τον κύριο Χόιε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η έκθεση, επενδύσεων, η έκθεση του κυρίου Μαρινέσκου αφορά ακριβώς